δώσουμε την εντολή. Παρατηρήσεις υπάρχουν, οπότε επικυρώνεται η εντολή της κυρίας Κάμεν και περνάμε στις ψηφοφορίες αρχής γενομένης από τις έκθεσεις Βιέφκα με απλουστευμένη διαδικασία για τη διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Με ονομαστική κλίση παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Μίλντερ. Για την κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών. Και πάλι με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Ροτ Μπέρεντ. Ε, για τα ειδικά προσωρινά μέτρα για την πρόσληση μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την ευκαιρία προσχώρηση τη Κροατία. Ποιο θέλει το λόγο, ο κύριο Λάντσμπαρκ. Είμαι υπέρ, αλλά δυστυχώ ε, δεν έχω μαζί μου την ηλεκτρονική κάρτα και για τι δύο εκθέσει. Ωραία, ονομαστική κλίση παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Ρόσμπαχ για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης. Διανατάσεις Ισχυρός που είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση Κρίστενσεν για τις ελευτικέ δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη Συμφωνία ελευτική Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνηση Ιδανία Με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση Κασίνη. Για το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε κατά τι εκλογέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από του πολίτε Ένωση που κατοικούν ένα κράτο μέρο το οποίο δεν είναι επίκοη. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση Colin Langen για την εφαρμογή της οδηγίας ε, που αφορά την καταναλωτική πίστη. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση για Ζωβιέτσκα. Για το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση Μποβέ. Για την ενημέρωση για τα γεωργικά προϊόντα και πρόθεσή τους. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, έκθεση Γκάλο για την εφαρμογή της οδηγίας για το δικαίωμα παρακολούθησης. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έκθεση Γκερέρο Σαλόμ για την τροποποίηση του άρθρου 70 του κανονισμού σχετικά με τις διοργανικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των νομοθετικών διαδικασιών. Ο εισηγητή ε, ζητά το λόγο, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λακωνικά δράτω με τι ευκαιρίε για να ευχαριστήσω τους σκιώδει εισηγητέ και του συντονιστέ τη Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων γιατί με υπομονή παρακολούθησαν ε, τις εργασίες και την δύσκολη διαδικασία έγκρισης αυτής της μεταρρύθμισης. Ζητήσα όμως το λόγο για να επισημάνω ότι η τροποποίηση του άρθρου 70 θα τεθεί σε ισχύ με το κανονικό σύστημα στις 10 Δεκεμβρίου, δηλαδή την πρώτη μέρα της επόμενης ε, περίοδου του Συνόδου της επόμενης Ολομέλειας και θα αρχίσει να ισχύει για τις νομοθετικές διαδικασίες για τις οποίες ε, η αρμόδια καθήλια επιτροπή δεν έχει υιοθετήσει, δεν έχει εγκρίνει ακόμη ούτε την ε, διαπραγματευτική εντολή, ούτε τη σύνθεση της ε, διαπραγματευτικής ομάδας. Καλώ το σημειώνουμε κύριε Γερέρο, ψηφίζουμε ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα... ζητώ συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Συγγνώμη, βιάστηκα, λέει η Πρόεδρος. Έχουμε τι ε, τροπολογίες όμω, 1, 4 και 6 μαζί. Θυμίζω ότι εδώ χρειάζεται ειδική πλειοψηφία υπέρ αυτών των τροπολογιών, 1, 4 και 6. Κατά. απόχέ, εγκρίνονται. Η τροπολογία παριθμών 3, το πρώτο τμήμα υπέρ, είναι κατά τμήματα, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμών 7 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία αριθμού 2 έχει καταπέσει συνεπώ και περνούμε ε, στι τροπολογίε 11 και 14 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται η τροπολογία 5 και η 18 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται η 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 και 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 και 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 8 σε δύο τμήματα τμήμα πρώτον υπέρ ε, κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτον υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 16 έχει καταπέσει. Η 10 υπέρ, κατά διστάζω λίγο, δεν σας βλέπω. Ονομαστική ψηφοφορία για τη 10 παρακαλώ, αρχίζει τώρα. Ε, στη δική πλειοψηφία θυμίζω εδώ. Πέρασε. Τις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται χρειαζόμασταν 377 ψήφους για να εγκριθεί. Η τροπολογία περισσότερων 16 ονομαστικά αρχίζει τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο της πρότασης. Εδώ αρκεί απλή πλειοψηφία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην επόμενη έκθεση του κυρίου Ήλτσεφ, ε, το, ε, τροποποίηση του άρθρου 181 του κανονισμού και του 182. Είναι και πάλι με ειδική πλειοψηφία υπέρ, κατά, απόχες, εγκριέται. Και η πρόταση, το σύνολο δηλαδή υπέρ, με απλή πλειοψηφία κατά, απόχες, εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην έκθεση του κυρίου Βαντεκάμπ. Έγκριση και εποπτεία της αγοράς δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων όπως και τετρακύκλων. 148 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, μπλοκ 1 μέχρι 147. Α, όχι, έχει καταπέσει, συγγνώμη. Ε, η τροποποιημένη πρόταση λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και το νομοθετικό ψήφισμα θα το ψηφίσουμε τώρα ονομαστικά. Αρχίζει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση του κυρίου Παντζέρη. Έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων. Έχουμε το πρώτο μπλοκ, η τροπολογία 320 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μπλοκ τροπολογιών λοιπόν καταπίπτει ε, η τροποποιημένη πρόταση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική κλίση αρχής του η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Έχουμε την έκθεση Τέρχο τώρα πληρωμές με κάρτα μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων. Για την παράγραφο 41 κατά τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές όμως. Σας παρακαλώ να το ελέγξουμε αυτό ηλεκτρονικά. Είναι το δεύτερο τμήμα. Αρχίζει της παραγράφου 41. Αρχίζει η ψηφοφορία. Και τελειώνει. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στην παράγραφο 43 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα της παράγραφου 43 υπέρ κατά αποχές και εδώ χρειάζεται παλήθευση αρχίζει το ηλεκτρονική ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 43 Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η έκθεση του κυρίου Ελχαντράουι, σκιώδης τραπεζικό σύστημα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έκθεση της κυρίας Κώστα, η προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Η παράγραφος 9, σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κυρία Κώστα, θέλετε το λόγο να πείτε κάτι ως εισηγήτρια παρακαλώ. Ναι, ένα λεπτό κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους αδέλφους ότι σήμερα είναι η 23η επέτειος της ε, σύμβασης για τα παιδιά του ΟΗΕ και θεωρώ ότι ο ψηφιακός κόσμος είναι το νέο όριο για την ε, προστασία των δικαιωμάτων ε, των παιδιών και των εφήβων. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής ε, Πολιτισμού, την συνάδελφο από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για τις Συνεργασίες της. Θεωρώ ότι σήμερα είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Κώστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το δεύτερο τμήμα της ΕΝΕΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 24, στα δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 34 υπέρ. Τσεκ. Καλά. Να ελέγξουμε την 32 τότε. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική επαλήθευση. Και τελειώνει. Εγκρίνεται. Παράγραφος 34. Ψήφι Π. Κατά. Αποχές. Ε, δεν είναι σαφές. Και εδώ παρακαλώ να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Σας παρακαλώ σηκώντε τα χέρια σας γιατί δεν σας βλέπω. 43 επέ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 επέ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη α σε τρία τμήματα τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη Δ, υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη και λατινικό ε, σε δύο τμήματα υπέρ. Κατά. Το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε ακόμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ελ λατινικό σε δύο τμήματα υπέρ. Το πρώτο. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας. Ερχόμαστε τώρα στην έκθεση του κυρίου Μπέκερ. Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Η τροπολογία 1. Ψήφι Π. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η παράγραφος 11. Υπέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η παράγραφος 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Nous allons maintenant nous arrêter pour la séance. Θα διακόψουμε τώρα για την πανηγυρική συνεδρίαση. le président haïtien. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αιτής. Un peu de contestation. S'ils insistent, on peut poursuivre. Bien, devant, devant, devant une telle protestation, je propose que nous... Μετά από αυτή την κατακραυγή ας συνεχίσουμε. Μια απόπειρα έκανα κι εγώ. Allons-y au travail, donc sur ce rapport Thyssen. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη δουλειά. Έκθεση Tyson, τροπολογία 1, ονομαστικά. Τώρα θα κλείσει η προσοχή η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 2. Επίσης με ονομαστική κλίση αρχής ψηφοφορία. Le vote Πέρας. Απορρίπτεται. Η παράγραφος 2. Μητροπολογία 3. Σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο με ονομαστική κλίση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Το δεύτερο τμήμα διανατάσεως υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 4, τμήμα πρώτον, ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία και τελειώνει. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα, διανατάσσεως χειρός υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία νέα σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο με ονομαστική κλίση αρχής ψηφοφορία και τελειώνει. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 10 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Πέρα. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 5, διανατάσσεως χειρός υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Με ονομαστική κλίση το παράρτημα αρχίζει τώρα η Ψηφοφορία. Δεν κρίνεται. Η τροπολογία 11 είπε Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 12 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Le vote est clos. Pérez. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 13, ονομαστική κλίση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Le vote est clos. Πέρας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη ΑΕ σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη CN. Με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ΣΕΠΕ. Ονομαστική κλίση. Ποιος θέλει το λόγο... Ε, για μετά, εντάξει. Ε, είμαστε στο ΣΥΠΗ με ονομαστική ψηφοφορία, αρχίζει τώρα. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Τάισεν. Έχουμε άλλη μια ψηφοφορία γρήγορα τελευταία για να σεβαστούμε το προσκεκλημένο μας. Η έκθεση του κυρίου Νόιζερ. Ε, μία ψηφοφορία είναι υπέρ, επί του συνόλου της εκθέσεως κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, Η κυρία Στριφλέ, ευχαριστώ Πρόεδρε, λυπούμε λίγο που η μερίσια διάταξη τροποποιήθηκε, διότι σήμερα υποδεχόμαστε πανηγυρική συνεδρίαση τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της ΑΕΤΗΣ. Θυμίζω, σας θυμίζω ότι η Ευρώπη είναι παριθμόν ένα ε, δωρητής παγκοσμίω ε, στην παροχή βοήθειας της ΑΕΤ και αν μη τι άλλο θα πρέπει με ευγενικό τρόπο να υποδεχθούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της ΑΕΤ. Λυπάμαι ειλικρινά που αλλάξατε την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ κυρία μου. Μα, μόλι έρχεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.